Colleagues, good morning. I think it's time to start. Καλημέρα σα, Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε άλλη μία προθεσμία της ψηφοφορίας. Καλώς ορίσατε. Έχουμε, ως συνήθω διερμηνία σε 17 γλώσσες. Συνήθω έχουμε παραπάνω είναι ουσιαστικά συνεδρίαση χωρίς έγγραφα και μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Έχουμε διαθέσιμα και τα πρακτικά της 30 Αυγούστου. Υιοθετούνταν δεν υπάρχουν σχόλια. Έχουμε μαζί μας σήμερα δύο προσώπους της ΜΠΟΣ δεξιά μου, ο κύριος Πίτερ Μπίζενμπαχ, διευθυντής του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων και τον ε, δόκτορα Μάικλ Κρούγκερ, ε, ανώτερο αντιπρόεδρο του Τμήματος Μηχανικής Συστημάτων ε, Diesel. Δύο εξαιρετικούς καλεσμένους και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπίζερμαχ για την εισαγωγή και θα περάσουμε στην ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Επιτροπή σας που κάλεσε την ΠΟΣ αυτή την ακρόαση και μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε στο σημαντικό σας έργο. Ονομάζομαι Πέτερ Μπίζενμπαχ, ε, είμαι επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων και Πολιτικής στην ΠΟΣ. Ε, μαζί μου είναι ο συνάδελφος Μίχαλ Κρούγκερ για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, ο οποίος είναι επικεφαλής ανάπτυξης συστημάτων diesel στην ΠΟΣ. Για να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι θα κάνω τα εισαγωγικά μου σχόλια και θα απαντήσω σε ερωτήσει σα στη μητρική μου γλώσσα. Και αφήστε με τώρα να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα της επιχείρησής μας. Η BOSS είναι μια ε, διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών με έδρα στη Στουτγκάρδη και πολύ ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ. Η BOS επενδύει σχεδόν 10% του κύκλου εργασιών της στην έρευνα και την ανάπτυξη και στην, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μάλιστα πάνω από το 10%. Η Bosch απασχολεί ε, ανά τον κόσμο από τους 375.000 ε, υπαλλήλους, σχεδόν 56.000 στην έρευνα και την ανάπτυξη σε 118 πόλεις. Τα περασμένα χρόνια. Είχαμε μάλιστα πάρει πολύ καλές θέσεις ε, στον κατάταξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ε, στις ε, δαπάνες για την ανάπτυξη. Η BOS δεν, ανήκει στο δεν είναι συγμένη στο χρηματιστήριο και ανήκει κατά 92% στο κοινοφαλές ίδρυμα Robert Bosch. Είμαστε σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας και Μάλιστα, όπως μας ρωτήσατε γραπτός, είμαστε ε, μία από τις τέσσερις ε, μεγαλύτερες εταιρείες προμηθευτές ε, ε κινητήρων, ε, μονάδων ελέγχου κινητήρα. Και όπως έχετε διαβάσει στον τύπο, είμαστε και ένας από τους προμηθευτές της Volkswagen πώς ε, προμηθεύει τη, τους ε, ψεκασμού, τις μονάδες ψεκασμού για τις δίλητρες μηχανές ε, diesel αλλά όχι ε, των υπολείπων. Το, για τους κινητήρες 1,6 και 1,8 ε, προμηθευτές είναι ανταγωνιστές μας. Εμείς προμηθεύουμε την αυτοκινητοβιομηχανία και υλικό και λογισμικό. Και εάν δούμε τις, τα, τελευταία τεστ κινητήρων diesel από τις Βρετανικές, Γαλλικές και Γερμανικές αρχές, η BOS ε, θα δούμε ότι προμήθευσε πολλές ε, εταιρείες και στις ε, δοκιμές 14 κινητήρων για το νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης 13 από τα 14 οχήματα πέρασαν το τεστ. Ε, τα τεστ αυτά έδειξαν επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη τεχνολογία για να μειωθούν οι εκπομπές σε οποιαδήποτε, υπό οποιαδήποτε συνθήκες οδήγησης. Γι' αυτό λοιπόν ε, περιμένουμε από εσά να μας ρωτήσετε για περισσότερες πληροφορίες, να ε, μάθετε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές, πώς ε, λειτουργούν τα συστήματα διαχείρισης εκπομπών. Είναι ένα περίπλοκο ε, σύστημα, περίπλοκες μηχανικές απαιτήσεις και μόνο ένα εξίσου περίπλοκο λογισμικό μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και ένα λογισμικό που θα τρέχει ε, χωρίς προβλήματα. Η BOS επίσης στηρίζει την υποχρέωση να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι εκπομπές και να δημοσιοποιηθούν οι να δημοσιοποιηθούν στις ε, αρχές οι προποθέσεις για την έγκριση τύπου. Ελπίζουμε λοιπόν η σημερινή μας παρουσία εδώ να συνεισφέρει σημαντικά στο έργο σας. Και θα ήθελα να πω άλλη μια φορά και να τονίσω ότι η τεχνολογία diesel μας επιτρέπει ε, να ε, έχουμε πολύ χαμηλές εκπομπές αυτό ισχύει και για τα σωματίδια και για το οξύδιο του αζότου. Και μέχρι τώρα όλες οι μελέτες από το ICCT μέχρι τις, ε, μέχρι τις εθνικές δοκιμές μας ε, δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα μπορούν να πιάσουν πάρα πολύ καλές τιμές όταν η ε, τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας εφαρμόζεται και η εισαγωγή των, ε, ε, των τεστ σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, πολύ σύντομα θα επιτρέψει σε όλα τα αυτοκίνητα, βενζινοκίνητα και δίζελ να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών. Η Bosch έχει στηρίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, την πρόταση για τεστ σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και ε, ακριβώς για να υπάρχει και η πολιτική αποδοχή και η αποδοχή από τους, ε, από τους πολίτες χρειάζεται ο κινητήρας να έχει χαμηλές εκπομπές. Γι' αυτό λοιπόν η, τα τεστ σε πραγματικές συνθήκες οδήγηση πιστεύω θα οδηγήσουν και πιστεύει και η εταιρεία μα πως θα οδηγήσουν ε, σε μια μεγαλύτερη ε, δημόσια αποδοχή. Για να μειωθούν ε, περισσότερο οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολύ αποδοτικ... έναν πολύ αποδοτικό κινητήρα ε, που θα έχει άμεσο ψεκασμό και στους κινητήρες δίζελ και βενζίνης. Η ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ηγείται της τεχνολογίας αυτής και η ΜΠΟΣ μόνο επενδύει κάθε χρόνο σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την... Για την για τον εξηλεκτρισμό ε, των κινητήρων. Έχουμε δει πως ε, αυτό είναι αναγκαίο για να μειωθούν ακόμα περισσότερο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, αν θέλουμε να ε, φτάσουμε αυτούς τους ε, πολύ φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις τεχνικές μας και τεχνολογικές μας δυνατότητες για να το καταφέρουμε και να διατηρήσουμε την ισχύ της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας. Ελπίζουμε λοιπόν με τη συνεισφορά μας να βοηθήσουμε το έργο της Επιτροπής σας και με χαρά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και μεγαλύτερη διαφάνεια. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι όπως γνωρίζετε και όπως διαβάζετε στα μέσα ενημέρωσης, οι κατηγορίες για την ε, παραποίηση, την αλλίωση του λογισμικού ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ε, ποινική εξέταση. Η ΜΠΟΣ ε, συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία και συνεργάζεται απόλυτα με τις αρμόδιες αρχές σε πολλές χώρες. Και ε, εξαιτία του ευαίσθητου αυτού λοιπόν ε, θέματος, επιτρέψτε μου να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για τις ε, διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα επίσης να ζητήσω την κατανόησή σας εάν εξαιτία αυτού δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε του περιεχομένου για, τη, για τις λεπτομέρειες ενώ σου βρίσκεται σε εξέλιξη μια, αυτή η δίκη. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι εμείς από τη στιγμή που ε, εμφανίστηκαν αυτές οι κατηγορίες οργανώσαμε στην ίδια μας την εταιρεία μια ε, εσωτερική έρευνα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόηση που θα δείξετε σε αυτά που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε μέχρι τώρα λόγω των νομικών περιορισμών και ε, είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι ερώτηση έχετε. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιζιμπάχ για τα εισαγωγικά σας ε, σχόλια αλλά και για τις ε, τελικές σας παρατηρήσεις. Γνωρίζουμε το θέμα αυτό, έχουμε και άλλες εταιρείε που προσκαλούμε στις ακροάσεις μας και είναι σε παρόμοια θέση. Τώρα, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, τον κύριο Σάλμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω σπανικά. Ευχαριστώ κύριε Κρούγκερ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, υπάρχουν διαφορές σε γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά την ε, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ε, στις εκδοχές ελαφρών οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά και την αμερικανική αγορά. Μπορούμε να πούμε ότι για κάθε όχημα, σε γενικές γραμμές και για κάθε μάρκα, υπάρχει μία, ε, ε, μία συγκεκριμένη λύση. Υπάρχουν διαφορετικές δηλαδή λύσεις, πολλές διαφορετικές λύσεις για κάθε ε, όχημα, για κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Ίσως αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει λοιπόν γιατί πρόκειψε και ανέκυψε το σκάνδαλο αυτό. Also das ist jetzt ziemlich spekulativ. Αυτές είναι οι κασίες. Δεν μπορώ να απαντήσω για το αν είναι αυτός ο λόγος. Δεν γνωρίζω. Ε, ε, Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Στην αξιολόγησή σας θα μπορούσατε να μας πείτε αν είναι δυνατόν τα αποτελέσματα του τεστ εκπομπών ε, θα μπορούσαν να παρεποιηθούν. Είναι δυνατόν να γίνει από τεχνική σκοπιά χωρίς να συμμετέχουν αυτά τα δύο τεχνικά στοιχεία. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα την ερώτησή σας. Θα μπορούσατε να ε, μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη σας, είναι δυνατόν από τεχνική σκοπιά τα αποτέλεσματα του τεστ εκπομπών να παραποιηθούν χωρίς να συμμετέχει ο προμηθευτής δηλαδή οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων. Ähm, ähm, Τα αποτελέσματα των εκπομπών είναι ε, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμείς. Ε, ένα ο, ε, καθήκον στα αυτά τα τεστ είναι να ε, μην ξεπεράσουν κάποια όρια. Ο κινητήρας ε, λοιπόν ευθύνεται για τα αποτελέσματα, ευθύνονται ατμοσφαιρικές συνθήκες, αντίσταση αέρα. Ε, είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Είναι πολλές οι συνθήκες που καθορίζουν τα αποτελέσματα των εκπομπών. Και ο, την επιστοποίηση δίνει ο κατασκευαστής του πρωτότυπου εξου, Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για το μέλλον με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα ξαναγίνουν τέτοια σκάνδαλα. Εσείς ε, πιστεύετε ότι λείπει κάτι και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να ζήσουμε αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Η νέα νομοθεσία περιέχει διάφορα καινούργια λοιπόν στοιχεία και εμείς θεωρούμε πως είναι τα σωστά μέτρα έτσι ώστε στο μέλλον ε, να διευκρινιστούν αυτά τα ασαφή σημεία στην ε, νομοθεσία και να αποκλειστούν τέτοιες ε, λοιπόν περιπτώσεις παρεπίσεις. Να σας ε, πω ότι για, τις, ε, για τα τέσσερα πραγματικές συνθήκες οδήγησης ο παλιός Επίτροπος Φερχόγγεν είχε ήδη ε, τοποθετηθεί πως ήταν ήδη γνωστή από τότε η διαφορά ανάμεσα στις, στα τέσσερα πραγματικές συνθήκες οδήγησης και στα, τεστ, εργαστηριακά τέστε. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και αυτή η απόφαση. Εμείς θεωρούμε πως είναι η, πολύ σωστή η απόφαση της εισαγωγής τέστε πραγματικές συνθήκες οδήγησης είναι φιλόδοξοι στόχοι και επίσης να πω ότι από τον Ιούνιο ήδη που ε, αποφασίστηκε αυτή η στρατηγική ε, να ε, συμπεριληφθεί και να αλλάξει την διαδικασία έγκρισης τύπου θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκέρμπραντι. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας που δέχτηκαν να περιβρίσκονται εδώ. Φυσικά κατανοώ απολύτως το γεγονός ότι δεν είστε σε θέση να αναφερθείτε σε ζητήματα που είναι υποποινική έρευνα, αν και είναι απογοητευτικό. Δύο ερωτήσεις για τη δική σας εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή και μπορούμε να περιμένουμε κάποια δημόσια έγγραφα, κάποια συνόψεις αφού θα έχει ολοκληρωθεί η έρευνά σας. Δεν είμαι νομικός, και δεν είμαι νομικός εκπρόσωπος της εταιρεία, αλλά οι έρευνες αυτές ε, άρχισαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και δεν μπορώ λοιπόν να σας πω πότε θα γίνει αυτό. Τώρα, ε, για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιμένετε τη ε, στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι έρευνες. Θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε σε ένα γραπτό σχόλιο που λάβαμε από έναν εμπειρογνώμονα λογισμικού που βρήκε μια συσκευή αναστολής ε, παραπίσης σε ένα αυτοκίνητο και απάντησε στην Επιτροπή μας έλεγε και θα παραθέσω στην περίπτωση της ακουστικής λειτουργίας, ε, δηλαδή που ανοιχνεύει ένα προφίλ οδήγησης ε, και καταλαβαίνουμε ότι εφαρμόστηκε από την ΠΟΣ που ουσιαστικά ε, βλέπει και ανοιχνεύει μία σχέση που έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν και το χρόνο. Όμως δεν έχει προγραμματιστεί από την ΠΟΣ κάτι παρά ε, δεδομένα που δεν είναι ακουστικά. Ποια είναι η αντίδρασή σας στη δήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μπορώ να πω πως ε, αυτό είναι ε, αντικείμενο των εξωτερικών ερευνών, όχι των εσωτερικών ερευνών στην εταιρεία μας. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Okay, well, that, that is quite disappointing. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είναι κάπως απογοητευτικό αυτό, γιατί θα μπορούσε να ειδωθεί μια γενική ερώτηση. Αλλά μήπως μπορείτε να δώσετε μια γενική απάντηση, όχι, πολυ... όχι επί συγκεκριμένων θυμάτων, αλλά μπορείτε να δώσετε κάποια γενική απάντηση, είναι δυνατόν. In θεωρητικά. Είναι ανάλογα την ερώτηση που μας κάνετε. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά θέματα. Θα προτιμούσα λοιπόν να μην απαντήσω. It was more about... Περισσότερο είχε να κάνει με το αν εσείς ως εταιρεία βάλατε στο λογισμικό αυτά τα dummy data, τα δεδομένα, που θα μπορούσαν ε, να συμπληρωθούν από έναν κατασκευαστή για να ε, ανοιχνεύσει αυτό αν έχει γίνει δοκιμή στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εσείς συμπεριλαμβάνετε μία λειτουργία για να μπορεί να ανοιχνευτεί ένας κύκλος δοκισμός που μπορεί στη συνέχεια να συμπληρωθεί από τον κατασκευαστή. Ωραία, σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν θα αναφερθούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε γενικέ γραμμές όμως, τεχνολογικά... Μπορούμε να πούμε πως... Ε, α, μάλλον θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρούγκερ να σας απαντήσει. Ναι, έχει ακουστεί νομίζω στην Επιτροπή από έναν συνάδελφο στην Volkswagen ότι χρειάζεται ένα τέτοιο ε, στοιχείο αναγνώριση στο λογισμικό γιατί υπάρχουν διάφορα συστήματα ε, βοήθεια, σταθερότητα για παράδειγμα και όταν εντοπιστεί, όταν ανοιχνευτεί ας πούμε από το λογισμικό ότι δεν κινούνται και οι τέσσερι τροχοί, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, τότε αυτό το σύστημα σταθερότητα πρέπει να απενεργοποιηθεί διότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η λειτουργία του αυτοκινήτου. Αυτό λοιπόν, αυτή η αναγνώριση για δεν είναι πρόβλημα, δεν αποτελεί πρόβλημα, δεν αποτελεί ε, παραποίηση. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, έχασα μερικά λεπτά. Δεν καταλαβαίνω αυτή την απάντηση. Γιατί χρειάζεστε λογισμικό που να αναχνεύει αν ένα αυτοκίνητο είναι σε δυναμομετρική εξέδρα. Ε, έχουμε άλλο λογισμικό για να δούμε αν είναι σε γκαράζ. Γιατί χρειάζεστε λογισμικό ε, για να ανοιχνεύει αν είναι σε κύκλο δοκιμών. Γιατί. Να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Όπως σας είπα, πώς να το πω καλύτερα, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, όταν βρίσκεστε λοιπόν σε αυτήν την ε, δυναμομετρική εξέδρια προσπαθούμε να προσωμιώσουμε συνθήκες οδήγησης σε, σε οδόστρωμα. Αυτό δεν είναι φυσικά το ίδιο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, υπάρχουν ε, παράγοντες ε, που αφορούν τη σταθερότητα του οδοστρώματος, αφορούν τα φρένα, αφορούν πολλά. Τώρα, όταν βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την εξέδρα. Μπορούν να γίνουν λάθη. Έτσι λοιπόν το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει αν κάτι δεν πάει καλά, αν υπάρχει κάποιο λάθος το οποίο δεν θα δώσει ένα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν το ε, λογισμικό να μπορεί να διαπιστώσει σε τι συνθήκες ε, οδηγεί το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω την ερώτησή μου στα γερμανικά, γιατί αυτές οι πολλές γλώσσες με μπερδεύουν. Στα αυτιά μου μπερδεύομαι. Λοιπόν, για να καταλάβω καλά, εσείς δεν είστε ε, OEM, εσείς είστε μόνο προμηθευτής. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Γκεμπράντι να το ρωτήσω αλλιώ. Εσείς μεταξύ άλλων προμηθεύετε την αυτοκινητοβιομηχανία με λογισμικό ή με μηχανήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μέτρηση εκπομπών. Ναι, ναι. Άρα, αυτό που εσείς προμηθεύετε είναι κάτι κλειστό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον ΟΗΕΜ ή είναι ένα ανοιχτό λογισμικό το οποίο μπορεί μετά κάποιος να αλλάξει. Λοιπόν, ναι, επί της ουσίας ε, το κόνσεπτ γύρω από τις εκπομπές αποτελείται από πολλά ε, υποσυστήματα. Ε, δηλαδή, το σύστημα ψεκασμού, για παράδειγμα, αποτελείται από πολλά, πολλά διαφορετικά συστατικά στοιχεία. Από μία αντλία, από ένα ψεκαστήρα, από διάφορα. Υπάρχει ένα σύστημα εξαερισμού, υπάρχει ένα σύστημα εξαερισμού, καταλύτες, φίλτρα, αισθητήρε. Έτσι λοιπόν βλέπετε πως υπάρχει μια σειρά από ε, εξαρτήματα. Υπάρχει ένας, δείτε το σαν ένα μπουφέ με πολλά διαφορετικά φαγητά και λοιπόν ο OEM διαλέγει αυτά που του αρέσουν για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σας απάντησα επαρκώς. Ναι, θα προσ... προσπαθήσω, προσπαθώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι μηχανικός. Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει ένας μπουφές. Υπάρχει η δυνατότητα ο OEM αυτόν τον μπουφέ να τον ε, τροποποιήσει έτσι, να διαλέξει τα κατάλληλα ας πούμε, φαγητά από τον μπουφέ έτσι, ώστε να ε, παραποιηθούν τα τεστ. Δεν μιλάω τώρα για τη Volkswagen, μιλάω γενικά. Ξέρω πως δεν μπορείτε να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Αλλά ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων μπορεί χωρίς τη δική σας βοήθεια να ε, παρακάμψει αυτά τα τεστ, να, να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. Ναι, δεν μπορώ να σας πω τώρα τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει με τα τεστ, αλλά όλο αυτό το σύστημα δεν το προμηθεύει μόνο η BOS. δεν, δεν είμαστε μόνο εμείς που τα φτιάχνουμε. Ο κατασκευαστή αυτή, αυτή, αυτές μέρες έχει πολλούς προμηθευτές. Όταν ας πούμε παίρνει ένα σύστημα ψεκασμού από την BOS, τότε ε, να είστε σίγουροι πως ε, δεν είναι όλα τα εξαρτήματα από εμάς. ε, ορισμένα μάλιστα ε, εξαρτήματα δεν τα κατασκευάζουμε καν. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο προμηθευτών και όλα αυτά συναρμολογούνται ε, για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτός δηλαδή στην ουσία για να επιστρέψω στο παράδειγμα με τον μπουφέ αυτός που ξέρει ε, τι τρώει είναι αυτός που έχει βάλει τα φαγητά στο πιάτο του. Εμείς δεν είμαστε αυτοί. Μάλιστα. Κύριος Κάριντς. Είπατε πως περίπου το 10% του κύκλου εργασιών σας πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όχι, όχι, όχι, όχι, να σας διορθώσω. Από τις, ε, από τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη, πάνω από το 59% πηγαίνει στην ε, έρευνα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και με, για τη Volkswagen τι γίνεται, τι ποσοστό είναι αυτό, ότι τι, ποια είναι τα νούμερα της συνεργασίας σας με τη Volkswagen. Αυτό σίγουρα δεν είναι μυστικό. Ε, δεν ξέρω προσωπικά το ακριβές νούμερο, αλλά μπορώ να επικοινωνήσω ε, ή να επικοινωνήσετε κι εσείς με τον ε, υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων της ΜΠΟΣ και θα σας δώσω τα στοιχεία αυτά. Uh, is... <laughs> Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν οι ερωτήσεις μας όταν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να απαντήσετε. Ε, θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους για τις ερωτήσεις, γιατί εγώ νομίζω δεν μπορώ να προχωρήσω. Κύριο Στάνς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δυστυχώς, ε, εγώ πρέπει να συνεχίσω στα αγγλικά γιατί και εμένα με μπερδεύουν οι πολλές γλώσσες στα αυτιά μου. Θα ήθελα να δούμε λίγο με το θέμα που ρωτήθηκε προηγουμένως. Ο σκοπός του σχεδιασμού του λογισμικού είπατε ότι είναι απαραίτητο να ανοιχνεύεται ε, το αυτοκίνητο όταν είναι σε δυναμομετρική εξέδρα. Ποια είναι τα σφάλματα, τα λάθη που ανοιχνεύεται έχουν να κάνουν με τις εκπομπές αυτές καθεαυτές, είναι μετρήσεις εκπομπών, μπορούμε να έχουμε σφαλμένα αποτελέσματα με αυτή την ανέχνευση όταν είναι σε εξέδρα. Υπάρχουν άλλα στοιχεία ασφαλείας που ανοιχνεύονται. Ποιος είναι ο σκοπός του σχεδιασμού αυτού του λογισμικού. Also, ähm, um Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας απαντήσω 100% σε αυτή την ερώτηση. Έχει να κάνει με, τη, με την ηλεκτρονική σταθερότητα, τον έλεγχο της ηλεκτρονικής σταθερότητας σε γενικέ γραμμές. Δηλαδή, σε κανονικές συνθήκες οδήγησης θέλουμε να μην ξεπεράσουμε κάποια όρια εκπομπών. Αυτό πρέπει να ε, γίνει όταν και οι τέσσερις τροχοί κινούνται. Όταν ας πούμε δύο από τους τέσσερις τροχούς δεν κινούνται, κάτι που συμβαίνει σε μια τέτοια δυναμομετρική εξέδρα, η οποία είναι εξέδρα προσωμείωσης. Και τονίζω το προσωμείωση, διότι η προσωμείωση δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό το, ε, αυτή η τεχνολογία λοιπόν μπορεί να εντοπίσει αυτά τα λάθη. Δηλαδή το ότι δεν λειτουργούν και οι τέσσερις τροχοί, βρίσκεται σε εξέδρα. Μπορεί δηλαδή να εντοπίσει κάποιο λάθος, αλλά ο σκοπός του δεν είναι να λιώσει αποτελέσματα, ο σκοπός του είναι να εντοπίσει το λάθος και να το διορθώσει. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος εξαντλητικός κατάλογος από το ποια λάθη είναι αυτά. Δηλαδή έχουμε σχεδιάσει αυτό το λογισμικό ας πούμε για να μην, ε, για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το λάθο. Αν δεν είναι εξαιρετικό ο κατάλογο αυτών των λαθών, ε, τότε αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι μα δίνει μεγάλη ευελιξία στο πώ το χρησιμοποιούμε. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα αυτό που με ρωτάτε. Πιστεύω πως ε, και ο, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Volkswagen αυτό είναι ότι η ο κινητήρας αναγνωρίζει ότι γίνεται ένα τεστ, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ε, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτή η αναγνώριση για να αλλοιώσουμε αποτελέσματα, να παραπείσουμε αποτελέσματα. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω στην ερώτησή σας ικανότητα να χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο χειραγώγησης είναι θέμα κανονισμών. Κατά την άποψή σας ποιος είναι υπεύθυνος να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει χειραγώγηση. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε να ρωτήσετε ποιος έδωσε την εντολή σε ποιον να γίνουν αυτές οι αλλοιώσεις, οι παραπίσεις. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ε, στο τέλος, το, το σύστημα ενός αυτοκινήτου, όπως σας είπα, συμπεριλαμβάνει διάφορα πράγματα. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Αυτό είναι και το, το νόημα της έγκρισης τύπου. Τώρα η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα του τεστ και στις πραγματικές εκπομπές ήταν κάτι που ήταν πάντα γνωστό. Δεν ήταν κάτι που αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε. Αλλά ε, και δεν μπορούν αυτά τα αποτελέσματα αυτά να είναι ολόιδια σε κάθε περίπτωση, σε κάθε δοκιμή. Δεν υπήρχε λοιπόν ποτέ κάποια ένδειξη πως έχει γίνει κάποια χειραγώγηση. Ε, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι αποτελέσματα των, ε, τεστ, των εργαστηριακών τεστ τα οποία πρέπει να επαναληφθούν σε πραγματικές συνθήκες. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Είπατε ότι είναι ευθύνη στο τέλος α, σχετικά με τη χειραγώγηση όχι, όχι την ε, ε, χειραγώγηση, αλλά αυτή την προσαρμογή, την customization που αναφέρατε. Εάν ένας πελάτης θέλει να προσαρμόσει ένα εξάρτημα, να το χρησιμοποιήσει με διαφορετικό τρόπο, ε, ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό, εσείς το κάνετε αυτό ή το επισκευάζετε το προϊόν. Okay. Είναι τεχνικό το ερώτημα, αλλά θα προσπαθήσω να το απαντήσω εγώ. Φυσικά, εμείς ως προμηθευτέ, είμαστε υπεύθυνοι για την ε, ένταξη όλων αυτών των εξαρτημάτων στο σύστημα. Για τα εξαρτήματα δηλαδή που προμηθεύουμε. Αυτή η διαδικασία λοιπόν συναρμολόγηση ε, συνδέεται με διάφορε άλλε εργασίε. εργασίες. Αλλά νομίζω πω εσεί ρωτάτε για την ε, για το ποιος έχει την ευθύνη για όλο το σύστημα οδήγησης, για όλο το σύστημα εκπομπών ενός αυτοκινήτου. Αυτό ε, δηλαδή, αυτή η ευθύνη δεν ε, είναι ευθύνη του, των επιμέρους προμηθευτών, είναι ευθύνη του τελικού αποτελέσματος, αφού είναι αποτέλεσμα συναρμολόγησης. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χένκελ. Κυρίες και κύριοι, για 25 χρόνια ήμουν στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της Bosch της Continental και Γι' αυτό λοιπόν, επειδή νομίζω πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, θα προτιμούσα να μην κάνω καμία ερώτηση στους εκπροσώπους της ε, ΜΠΟΣ. Ε, ε, θα μιλήσω σουηδικά για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, που προσπαθείτε τουλάχιστον να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα να προσπαθήσω να υιοθετήσω μια κάπως διαφορετική προοπτική σε σχέση με τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Εάν ένας κατασκευαστής σας παραγγείλει εξαρτήματα για το όχημά του, έχετε κάποιον έλεγχο για να ελέγξετε ότι τα εξαρτήματα που παραδίδεται ε, συμμορφώνονται ε, προς ε, τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν. Ναι, υπάρχει διαχείριση ποιότητας, υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία και σε εμά και στην πόση η οποία διασφαλίζει ότι τα επιμέρους εξαρτήματα ε, πληρούν τις ε, προϋποθέσεις. Ε, τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι γενικότερος έλεγχος ποιότητας για όλα, αλλά αυτό που σας είπα το έχουμε. Αυτή ήταν μια καλή απάντηση, γιατί προσπαθούμε εδώ να δούμε τι συνέβη και εσείς ε, ως προμηθευτής εξαρτημάτων είστε σημαντικό μέρος ε, της αλυσίδας και όταν ε, κατασκευάζετε εξαρτήματα που περιλαμβάνουν λογισμικό τότε αφήνετε επίτηδες χώρο έτσι ώστε ο κατασκευαστής πρωτότυπου εξαρτησμού να κάνει προσαρμογές στο σύστημα ή προσπαθείτε να το κλείσετε έτσι ώστε το εξάρτημα που παραδίδετε εσείς στον κατασκευαστή να είναι το τελικό προϊόν και να μην μπορεί να προσαρμοστεί εκτός αν ο ίδιος ο κατασκευαστής κάνει τεράστια τεχνική προσπάθεια. Έτσι όπως κάνατε την ερώτηση δεν μπορώ να την απαντήσω 100%. Ε, Το λογισμικό αποτελείται από πολλά στοιχεία. Υπάρχει δηλαδή ε, καταρχάς η πλατφόρμα η οποία έχει την αρμοδιότητα να συναρμολογήσει τα διάφορα εξαρτήματα. Τώρα, αν για παράδειγμα θέλετε ένα συγκεκριμένο ε, σύστημα ψεκασμού, πρέπει να προσθέσετε αυτό το σύστημα. Ε, υπάρχει ένα σύστημα πίεσης για παράδειγμα. Πρέπει δηλαδή κάποιος ε, όταν ε, θέλει να θέσει λειτουργία αυτό το σύστημα να πατήσει το αντίστοιχο κουμπί ας πούμε. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες σε αυτήν την πλατφόρμα. Αλλά υπάρχει λοιπόν αυτό το βασικό λογισμικό, η πλατφόρμα, το οποίο δεν το κάνει η BOSS, το κάνουν οι ανταγωνιστές της BOSS. Μετά υπάρχουν συγκεκριμένα εξαρτήματα τα οποία μας ζητάει ο πελάτης. Ο πελάτης για παράδειγμα μπορεί να μας ζητήσει κάποια, κάποια στοιχεία ε, που θέλει αυτός να περιέχει το λογισμικό. Διάφορα ε, σε γενικές γραμμές, λοιπόν, όταν μας ζητούν κάτι, μπορούμε να ξέρουμε περίπου γιατί το θέλει, αλλά δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα, ένα είδος μαύρου κουτιού που ε, υπάρχει σε αυτό το λογισμικό. Τώρα, τα συστήμα, το λογισμικό αυτό όπως το καταλαβαίνετε εσείς, είναι μία συνεργασία ανάμεσα σε λειτουργίες και σε δεδομένα που, ε, που, τα, τροφο, τα δίνει κάποιος αυτό το λογισμικό. Ε, αυτά όμως σε γενικέ γραμμές τα, προ, τα προμηθεύει ο κατασκευαστής του πρωτότυπου εξοπλισμού. Αυτός αποφασίζει τι θέλει να κάνει με το λογισμικό. Ε, Ευχαριστώ. Ακόμα δύο μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη... σχετικά με αριθμούς πόσα οχήματα δίζελ στην Ευρώπη κυκλοφορούν με ελέγχους της Bosch, χοντρικά πόσα οχήματα και άλλο ερώτημα συμπληρωματικό σαν όσα είπατε προηγουμένως. Αισθάνεστε ασφαλείς, σίγουροι για τα προϊόντα που παραδίδετε στον κατασκευαστή. Είσαστε βέβαιοι ότι τα εξαρμήματα που παραδίδετε είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους ε, τα νόμους ή υπήρξε κάποιο σφάλμα, υπήρξε κάποια παρέκκληση ε, και μήπως ο κατασκευαστές χειραγώγησε ή παραποίησε ορισμένα πράγματα εκ των υστέρων. Δεν ξέρουμε ακριβώ τον ακριβή αριθμό των δίζελ αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν τον έχουμε ε, προχειρώσει. Μα συγχωρείτε λοιπόν, ε, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλέ γενιέ δίζελ. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό έτσι αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια μπορούμε να σα ε, δώσουμε γραπτό αυτή την απάντηση αργότερα. Να σα πούμε τον ακριβή αριθμό των δίζελ αυτοκινήτων που ρωτήσατε. Τώρα, Τώρα, μα ρωτήσατε δηλαδή πόσο αυτοκίνητα diesel υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με εξαρτήματα δικά μα, τη BOS. Να σα πω ότι αυτά τα εξαρτήματα, τώρα για το όλο σκέλος της ερώτησής σας, ε, είναι σωστά. Λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Ε, πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης, είναι καθόλου νόμιμα και στην διαδικασία ελέγχου ποιότητας στην ΠΟΣ που σας ε, περιέγραψε ο κύριος Κρούγκερ δεν ακολουθούμε την αρχή της τεχνικής, ποιο... ποιότητας αλλά την αρχή του... της ε, νομιμότητας. Πρέπει δηλαδή εμείς, και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε, να ε, δίνουμε στην αγορά εξαρτήματα τα οποία είναι νόμιμα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, πληρούν τους κανόνες. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να αλλάξει την λειτουργία, το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας δεν μπορώ να το απαντήσω. Θα προτιμούσα λοιπόν να μην το απαντήσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της ΜΠΟΣ για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Αν και φοβάμαι ότι οι απαντήσεις ε, δεν μας διαφωτίζουν και πολύ, δεν διασκεδάζουν τις αμφιβολίες που έχουμε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Στις γραπτές σας απαντήσεις, εσείς αρνείστε οποιαδήποτε ευθύνη στην τελική χρήση του λογισμικού αλλίωση των εκπομπών. Παρ' όλα αυτά, δέχεστε ότι η δημιουργία αυτή τη τεχνολογία ε, γίνεται από τον ε, κατασκευαστή και επίση ε, δώσατε σημαντικά ποσά εναντί των πιθανών κυρώσεων που μπορεί να επιβληθούν από τα δικαστήρια και αν ε, ε, δούμε κάποια μέλη που έχουν στελθεί στην Volkswagen που αναφέρονται στην παραπίση και στη χειραγώγηση αυτού του λογισμικού ε, αυτό είναι βέβαιο ότι έχει γίνει τα παρελθόντα χρόνια. Μπορείτε να μας σχολιάσετε αυτά που υπονοούν ότι πως ήξερε ότι η Volkswagen χρησιμοποιούσε αυτό το λογισμικό για να προβεί στην παραποίηση που ανακαλύφθηκε από τις Αμερικανικές Αρχές. Καταλαβαίνω την ερώτηση, καταλαβαίνω και τον ενδιαφέρον σας, αλλά παρακαλώ να δείξετε κατανόηση, διότι αυτό που με ρωτάτε είναι ε, αντικείμενο και της εσωτερικής έρευνας και των εξωτερικών ε, ποινικών ερευνών, γι' αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Ε, Η Bosch ε, προμηθεύει διάφορους κατασκευαστές και των οποίων οι πραγματικές εκπομπές ξεπερνούσαν τα όρια που έχουν τεθεί στη νομοθεσία μέσω διάφορων μηχανισμών, μέσω δημοτικών παρατηρητών. Εγώ θα ήθελα να δω ε, ότι δεδομένου της προηγούμενης απάντησής σας ε, που λέτε ότι υπήρχε αυτό το λογισμικό σε μια σειρά εξαρτημάτων, θέλω να ρωτήσω αν ήταν απαραίτητο αυτό το λογισμικό έτσι ώστε τα αυτοκίνητα να μπορούν να παράγουν εκπομπές ε, που να είναι συμβατές ε, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε συνθήκες δοκιμών. Προσπαθήσω να απαντήσω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας. Φυσικά κάθε κινητήρα χρειάζεται και ένα λογισμικό για τον κινητήρα. Είναι βασικό συστατικό στοιχείο για όλη την ε, στρατηγική μέτρηση εκπομπών και μείωση εκπομπών. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά την ερώτησή σας, με ρωτάτε εάν κάθε κινητήρας ε, χρειάζεται αυτόν τον, αυτή τη μονάδα ελέγχου κινητήρα. Ε, ναι, εμείς είμαστε ένας από τους ε, τρεις μεγάλους προμηθευτές ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κυβωτίου ταχυτήτων ε, για παράδειγμα, της Volkswagen. Αυτό ας πούμε το έχουμε προμηθεύσει εμείς. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ίσως σας βοηθήσει αυτό που θα πω. Από ό,τι Καταλαβαίνω. Μιλάτε για ένα λογισμικό το οποίο τελείωσε, το φτιάξαμε, κλείνει, το δίνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Φανταστείτε, θα τα πω έτσι πολύ απλά τα πράγματα, ότι παίρνετε ένα αρχείο Excel και πρέπει να το... Πρέπει να βάλετε στοιχεία για να δουλέψει το πρόγραμμα. Κάπως έτσι γίνεται και με αυτό το λογισμικό. Πρέπει δηλαδή να τροφοδοτηθεί με δεδομένα και μετά θα γίνει κάτι. Αυτό δηλαδή το λογισμικό που λέτε εσείς δεν υπάρχει. Eh, Θα ήθελα να μου πείτε επίσης αν κάποια στιγμή ε, ουσιαστικά εξετάσατε τις αποκλίσεις ε, μεταξύ των πραγματικών εκπομπών και των υποτιθέμενων εκπομπών των αυτοκινήτων που εσείς προμηθεύετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις Εθνικές Αρχές ε, προκειμένου ε, να γίνει σεβαστή η νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τις εκπομπές των οξυδίων του αζότου. Μπορώ να πω ότι η ΜΠΟΣ σε αυτήν την ε, διαδικασία φυσικά και συμμετέχει. Συμμετέχει στην ε, διαδικασία, συμμετέχει στην ε, προσπάθεια για βελτίωση της νομοθεσίας. Έχουμε συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις εθνικές αρχές. προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τους, τις ενώσεις αυτοκινήτων, ενώσεις προμηθευτών, κατασκευαστών, συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνονται διαβουλεύσεις, αυτές έχουν δημοσιευτεί και όλα. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτά και επίσης βρισκόμαστε σε συνομιλίες όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και μάλλα με όλες τις αρμόδιες αρχές και, με, και επίσης βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με τους αρμόδιους ηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να έχουμε στη, να αναδώσουμε ε, όλα τα αναγκαία στοιχεία στη διάθεση των ε, αρμόδιων φορέων για να μπορέσουμε έτσι να ε, βοηθήσουμε στο έργο αυτό. Βοηθάμε λοιπόν, συνεργαζόμαστε πολλές φορές μας καλούν και καλούν δικούς μας επιρρογνώμονες ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τους δείξουμε ε, τις τελευταίες εξελίξεις, να δούμε και συνεργαζόμαστε σε γενικέ γραμμές για την νομοθεσία. Ο κ. Σέικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Δεν είναι εύκολο να θέτει κανείς ερωτήσεις, ε, γιατί πολύ γρήγορα μπαίνει κανεί σε τα νερά, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιε πιο γενικέ ερωτήσει, τι οποίε μπορείτε να απαντήσετε. Στην εισαγωγική σα δήλωση είπατε ότι οι μονάδε ελέγχου εκπομπών είναι διαθέσιμοι σε όλε τι συνθήκε οδήγηση και ότι σε όλε τι συνθήκε οδήγηση μπορείτε ουσιαστικά να έχετε ένα σταθερό όριο. Σωστό είναι αυτό ich glaube, Νομίζω πως αυτή τη στιγμή με ρωτάτε τι γίνεται στα τεστ, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό ε, δεν είναι καινούριο. αυτή η τεχνολογία, να σας πω, πώς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου για, την, ε, για τις, ε, τις εκπομπές υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν και διαφορές ανάλογα με τον κατασκευαστή, μειώνονται, μη, ε, οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές, δηλαδή αλλάζει η θερμοκρασία, αλλάζουν οι εκπομπές. Όταν ας πούμε ένα αυτοκίνητο οδηγεί σε κίνηση, αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, αυξάνονται οι εκπομπές, τότε πρέπει να γίνει μια ε, επανεπεξεργασία. Υπάρχει, υπάρχει τεράστια διαφορά λοιπόν ε, στον τρόπο της επεξεργασίας. Ε, διαφορές που έχουν να κάνουν με την πίεση όπως σας είπα. Έπειτα, τι θα γίνει με αυτές, ε, με αυτές τις ε, εκπομπές, με την εξάτμιση, πού θα πάει το αέριο, πώς θα ανακυκλωθεί, πού θα μπει αυτός ο ε, αεραγωγός, πού θα μπει το μηχάνημα για την ψήξη του αερίου αν δείτε ας πούμε ε, τι γίνεται στον χώρο αυτό, αν δείτε ας πούμε την καινούργια, το καινούργιο σύστημα που χρησιμοποιεί η Mercedes, θα δείτε ότι έχει κάνει άλματα η τεχνολογική πρόοδος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζει και εξελίζεται συνέχεια. Οι συνάδελφοι στη Volkswagen μας είχαν βάλει ένα όριο θερμοκρασίας μείων 25 βαθμών. Ε, αλλά στο μέλλον να είστε σίγουροι πως θα βελτιωθούν πάρα πολύ τα πράγματα. Θα προχωρήσει η τεχνολογία. Κοιτάξτε, ακούγεται ότι τεχνικά είναι δυνατό να μείνουμε εντός των ορίων και μάλιστα ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Επομένως, να κάνω μία ακόμη ερώτηση, γιατί αναφερθήκατε στις ψυχές συνθήκες. Θα ήταν ε, λογικό ότι στις ψυχρές ε, συνθήκες ε, η μονάδα έχουν κινητήρια να μην λειτουργεί πλήρως και θα ήταν οι οι εκπομπές ε, αν έχουμε θερμές συνθήκες ε, στην αρχή, στην έναρξη, δεν είναι. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένας καταλήτης χρειάζεται ένα συγκεκριμένο όριο θερμοκρασίας για να λειτουργήσει. Χημεία είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, έχει, αυτό λοιπόν, ε, αυτή λοιπόν είναι η απάντηση. Τώρα, όταν το πρωί, ας πούμε, σε μια κρύα μέρα, βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητό μου και έχει μείνει όλο το βράδυ στο κρύο, ε, είναι, ε, άλλο το πράγμα. Εξαρτάται όμω. Αν πάρω το αυτοκίνητο που έχει μείνει όλη τη μέρα στο κρύο, το βράδυ στο κρύο για να πάω στο φούρνο, φυσικά και εκπομπέ θα είναι πολύ μεγαλύτερε από ότι αν πάω να κάνω πολλά χιλιόμετρα για να πάω στη δουλειά μου, πούμε, σε μισή ώρα απόσταση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που επηρεάζουν το ε, όριο των εκπομπών και υπάρχουν και διάφορε συνθήκε οι οποίε μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τι εκπομπέ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για αυτή την ψυχρή έναρξη. Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχουμε καιρό. Όταν το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών στα 58 από τα 63 αυτοκίνητα βλέπει ότι τα πάνε καλύτερα τα αυτοκίνητα όταν έχουν ψυχρή έναρξη, παραθερμή έναρξη, μόνο πραγματική εξήγηση μπορεί να βρεθεί στο λογισμικό, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις με διαφορετικό τρόπο. Αυτές είναι οι εικασίες πρέπει να σας πω. Σας είπα το παράδειγμα με τον καταλήτη, αλλά αυτή η ερώτηση νομίζω πως ε, καλύτερα πρέπει να απαντηθεί από έναν συνάδελφο κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού. Εγώ δεν μπορώ να σας την απαντήσω. Ε, σωστά τα λέτε για τον καταλήτη, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο καταλήτης είναι ένα μόνο στοιχείο από το όλο σύστημα ελέγχου των εκπομπών. Μάλιστα, τότε θα εξάγω τα δικά μου συμπεράσματα. Και μια τελική ερώτηση, γιατί ήταν μακρύ και λύση απάντηση. Κάποιο κράτο μέλος σας έδωσε οποιαδήποτε ένδειξη ότι το λογισμικό ε, που μειώνει τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου των εκπομπών μπορεί να γίνει νόμιμα μόνο αν γίνει σε εργαστήριο παρά σε εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή είχατε κάποια τέτοια ένδειξη ότι αυτό απαιτείται σε εγκαταστάσεις δοκιμών. No, das ist mir nicht bekannt. Όχι, όχι, δεν το ξέρω κάτι τέτοιο. Mrs. Evie. Sì, grazie. Eh, ε, buon... Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Να σας ρωτήσω και ε, από Οτι η Bosch ε, θα είχε εντοπίσει τη Volkswagen ότι ε, αυτό το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στα αυτοκίνητα που είχε σε εμπορία θα μπορούσε να είναι παράνομο. Υπάρχει μια τεκμηρίωση της δήλωσή σας. Δηλαδή, εσείς είχατε ζητήσει ή λάβατε ε, ουσιαστικά ε, την ε, δυνατότητα να, προ... να μπορέσετε να υπερασπίσετε τα δικά σας συμφέροντα αν χρησιμοποιούνταν αυτός ο μηχανισμός, όπως φαίνεται ότι έγινε τελικά στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνω την ερώτηση, κατανοώ το ενδιαφέρον σας, όμως ε, λυπάμαι γιατί αυτό ακριβώς είναι κάτι που βρίσκεται σε αυτήν την ε, διαδικασία έρευνα. Είναι αντικείμενο ποινικών ερευνών. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Το φαντάζομαι. Σημειώνω το γεγονό ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε. Επομένω, θέλω να σα ρωτήσω. Από όσα είπατε μέχρι τώρα και βάσει και τη εμπειρία σα, πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν να ελοποιηθεί ένα λογισμικό ή ένα συνδυασμό λογισμικού και άλλων μηχανισμών, άλλων διατάξεων που να είναι σε θέση να προετοιμάσουν τα αυτοκίνητα για τα νέα τεστ, για τα νέα πέμψε, δηλαδή με φορητά συστήματα και να μπορούν να εγγυηθούν ε, ουσιαστικά τις καλύτερες επιδόσεις του κινητήρα με τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές. Also, ähm, da wage äh, ναι, θα τολμήσω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες, ε, πάντα υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι διασφάλισης αυτού. Τώρα το PEM στο φορητό σύστημα, όταν το, όταν το βάζουμε στο αυτοκίνητο, πρέπει ε, να λαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες από το όχημα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κάνει τις μετρήσεις σωστά. Χρειάζεται συγκεκριμένα δεδομένα για τις συνθήκες οδήγησης σε ε, οδόστρωμα, για παράδειγμα πού ακριβώς οδηγεί, τι, πώς είναι ο δρόμος ε, και μετριέται, μετράει σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα χρειάζεται για να μην οδηγηθούμε σε αυτές τις περιπτώσει που περιγράψατε εσείς. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ. Ελπίζουμε να μπορούσαν να λειτουργήσουν τα συστήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, έχω μια ερώτηση για το μέλλον και για να παρέμβουμε και με τις ισχύουσε νομοθεσίας για να την βελτιώσουμε, αν είναι δυνατόν. Κατά την έποψή σας, αρκεί να ζητήσουμε από τους προμηθευτές των κατασκευαστών να καταγγέλουν την παρουσία μηχανισμών διατάξεων παρεμβολής ε, στην φάση της έγκρισης τύπου. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να λένε λεπτομερώς, να δίνουν λεπτομερώς τις τεχνικές πληροφορίες ε, για τα λογισμικά που θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην αρχή ελέγχου έτσι ώστε αυτή να μπορεί να δει στη συνέχεια πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το software για να μπορεί να το ελέγξει πλήρως και για να μην ε, χρειάζεται να εμπιστεύεται την απλή δήλωση. Aus Regulierungssicht ist für die η έγκριση ενός οχήματος ε, είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Ε, από αυτό το θέμα έκμησης ε, τώρα όσον αφορά τη στρατηγική εκπομπών σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό ο οποίος ε, πρόκειται να δημοσιευθεί ένα τμήμα του λογισμικού πρέπει να, κοινο, να κοινοποιείται αυτό το AIS έχει ήδη ε, εγκριθεί τον Ιούνιο. Τώρα η ευθύνη για την έγκριση οχημάτων, για την έγκριση τύπου οχημάτων, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού, αλλά και ε, άλλων πραγματών. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Πρέτσελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση για ε, μία γραπτή απάντηση που δώσατε για την ερώτηση 2. Αν κατάλαβα καλά, λέτε πως έχετε δικές σας ποσοστώσεις, δικές σας προδιαγραφές, όμως εφαρμόζετε και τις ε, χρησιμοποιείτε και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού του OEM. Όμως όταν κάποιος δεν ξέρει αυτές τις προδιαγραφές του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού, τι ακριβώς συμβαίνει, τι προβλέπετε. Αλλάζει εκεί το πράγμα ή ε, ποιος ξέρει τι, τι, τι εννοείται δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε. Τι, είναι, αν είναι τεχνικής φύσης το ερώτημα να σας το απαντήσω. Όχι εννοώ για τη Volkswagen. Τι, αν εννοείται τη Volkswagen δεν μπορώ να σας απαντήσω, όμως μπορώ να σας απαντήσω γενικότερα. Ωραία. Γενικότερα, η γενική απάντηση είναι κάτι που έχουμε λάβει γραπτό. Σε μένα με ενδιαφέρει τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκτός Ωραία, θα κάνω μια γενική ερώτηση τότε. Όταν εσείς χρησιμοποιείτε αυτές τις ε, προδιαγραφές του κατασκευαστή πρωτοτύπου εξοπλισμού, δεν γνωρίζετε ποια δεδομένα στο τέλος ε, θα ε, χρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να αναγνωρίσετε όμως ότι κάποια δεδομένα είναι εκεί τα οποία δεν είναι αναγκαία ας πούμε για την ε, ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δυστυχώς πρέπει να πω αλλά θα σας πω το εξής. Δείτε για παράδειγμα πόσα, από πόσα δεδομένα αποτελείται ένα λογισμικό. Υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση 35.000 διαφορετικά ε, επιμέρους ε, δεδομένα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ, κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Όταν κάποιος δεν έχει το αυτοκίνητο μπροστά του είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει τι γίνεται ακριβώς. Γι' αυτό είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δύσκολα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και δεν θέλω να αποκλείσω ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις ε, που αυτό συμβαίνει. Είναι η εξαίρεση όμως, αυτό θα σας πω. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ε, δεν μπορείτε να μας απαντήσετε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά θα μπορούσε. Τώρα, στο τμήμα ανάπτυξη προϊόντων. μας είπατε πως ασχολείστε πάρα πολύ με την ποιότητα, πως ασχολείται και με την ποιότητα, ποιότητα ε, τι γίνεται όμως με την ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη όταν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, βασισμένοι σε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχουμε αυτή την εσωτερική έρευνα και βρίσκεται να εξελίξει όπως σας είπα. Μπορείτε να μας πείτε Ποιοι άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ε, χρησιμοποιούν προϊόντα της Bosch, εκτός από τη Volkswagen, για τα συγκεκριμένα οχήματα. Ε, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειε, όμως νομίζω πως σχεδόν όλους τους κατασκευαστές. Μάλιστα, μετά από το σκάνδαλο με τη Volkswagen υπήρξε εσωτερική έρευνα και για τους άλλους κατασκευαστές. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί αυτή τη στιγμή ε, αυτό που ρωτάτε είναι αντικείμενο των εσωτερικών μας ερευνών. Ωραία. Τότε φοβάμαι ότι και οι επόμενες ερωτήσεις μου δεν θα μπορούν να απαντηθούν για τους ίδιους λόγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρούγκερ, κύριε Βίζενπαχ που ήρθατε. Γνωρίζουμε ο... Γνωρίζετε ότι αυτή εδώ είναι μια εξεταστική επιτροπή και Κύριε Μπίζενμπαχ, μας ε, είπατε πως ε, δυστυχώς είστε περιορισμένος από τις εσωτερικές έρευνες και δεν μπορείτε να μας απαντήσετε στις περισσότερες ερωτήσεις. Ε, οι ποινικέ έρευνες αφορούν τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά οι εσωτερικές έρευνες γίνονται στην εταιρεία σας. Ε, πότε ε, μπορείτε να μας πείτε, ε, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εσωτερικές έρευνες. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτή την ερώτηση την απάντησα νωρίτερα. Ήταν ερώτηση μια συναδέλφου. Τώρα το πότε θα ολοκληρωθούν οι εσωτερικές έρευνες δεν μπορώ να σας το πω. Αυτή είναι μια διαδικασία ε, που κρατά πολύ καιρό. Δεν μπορώ λοιπόν να προβλέψω πότε θα ολοκληρωθεί. Τώρα ερώτηση για, την την ποινη... για τις ποινικέ έρευνες. Ε, αυτό με ρωτήσατε έτσι, πότε θα ολοκληρωθούν οι ποινικέ έρευνες. Ποιος διεξάγει τις εξωτερικές ανεξάρτητες έρευνες. Ξέρω πως στη Volkswagen ε, υπάρχει ε, ένα ανεξάρτητο φορέα που διεξάγει τι έρευνες. Ε, κοιτάξτε, έχουμε πρόβλημα. Σας κάνουμε ερωτήσεις, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Χαμένος χρόνος και για μας και για σας. Ε, δηλαδή, τι, πρέπει δηλαδή να ξανασυναντηθούμε σε έξι μήνες και να ελπίζουμε πως θα, θα έχετε κάποιε απαντήσεις. Δεν μπορείτε να μας πείτε τίποτα για τις ε, έρευνες, αλλά τέλος πάντων, 11.2, ε, ερώτηση 11.2. Μας απαντήσατε ότι τα όρια ότι οι προϋποθέσεις για το λογισμικό ορίζονται από τους κατασκευαστές. Όμως, ε, τι γίνεται με τον έλεγχο ποιότητας ε, νομικά, τι γίνεται με την νομική ευθύνη. Μας είπατε ότι υπάρχει μια γενικότερη πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να μπουν τα συστατικά που έχει ε, ζητήσει ο πελάτης και μετά τι γίνεται νομικά, δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη σε αυτό. Από πότε εσείς δεν έχετε πλέον ευθύνη για το τι γίνεται πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Υπάρχει δηλαδή κάποιο έγγραφο, κάποια σύμβαση που να λέει ότι από αυτό το σημείο και μετά εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για το τι γίνεται με το λογισμικό. Πολύ να απαντήσω στην ερώτησή σας, όμως δεν είμαι δυστυχώς νομικός και δεν μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα είναι σωστή απάντηση που θα σας δώσω. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω. Αλλά θα το κάνουμε γραπτός. Οι νομικές υπηρεσίες σας θα απαντήσουν σε αυτό. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν την γραπτή σας απάντηση. Μας είπατε πως παρακολουθήσατε και την προηγούμενη ακρόαση με τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι γραπτός μας είπαν ότι ε, πάνω από ε, ότι εκατοντάδες μάλλον μηχανικοί συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία της ε, συναρμολόγησης της αυτολογισμικού. Αλλά μετά ακούστηκαν, ακούστηκε ένας τελείως διαφορετικός αριθμός, ακούστηκαν πολύ λίγοι ας πούμε μηχανικοί. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτό το, αυτό το, το νούμερο που είπαν. Θεωρείτε ρεαλιστικό αυτό το νούμερο. Ε, κοιτάξτε, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, είπαν έναν αριθμό. Δεν μπορώ να, να αξιολογήσω αν αυτός ο αριθμός ε, ισχύει ή όχι, αλλά γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες. Έχει να κάνει με μια σύνθετη διαδικασία που πρέπει να αξιολογήσουν και να ανακατασκευάσουν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν για το αν μπορεί να ξέρει ένας μηχανικός όλα αυτά τα πράγματα, αν λίγοι μηχανικοί μπορούσαν να ε, κάνουν αυτό το πράγμα στο λογισμικό, αλλά όπως σας είπα, αυτά είναι αντικείμενα των εσωτερικών ερευνών μας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η δημιουργία, η συναρμολόγηση, ε, ο σχεδιασμός ενός, ε, μιας μονάδας ελέγχου κινητήρα είναι ένα αντικείμενο, είναι ένα έρευνας και ανάπτυξης πάρα πολλών ετών. Περνάνε πάρα πολλά χρόνια από το σχεδιασμό μια, ενός κινητήρα μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά σαν αυτοκίνητο. Ωραία, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Όταν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κατασκευάσουμε έναν κινητήρα καύση, αυτό δεν είναι μια δουλειά που την κάνουν δύο-τρει άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ε, που συμμετέχουν. Χρειάζεται πάρα πολύ ε, γνώση, μεγάλη τεχνολογία. Το λογισμικό από μόνο του δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν, υπάρχει το λογισμικό, υπάρχουν τα συστατικά στοιχεία του λογισμικού, υπάρχει στην μονάδα ελέγχου το σύστημα ψεκασμού, το σύστημα ανακύκλωσης των ε, εκπομπών, υπάρχουν διάφορα ψήξη. Υπάρχει ένας μεγάλος, μεγάλος λοιπόν αριθμός ε, μηχανικών, ο οποίος ασχολείται με αυτό το μικρό εξάρτημα. Ευχαριστώ πολύ. προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά παρόλο που είναι δύσκολο για μένα. Για να βεβαιωθώ ότι καταλαβαίνω τη δομή. Εσείς είστε προμηθευτές εξαρτημάτων ε, για τους κατασκευαστές πρωτοτύπων εξοπλισμών και επίσης κατασκευάζετε και εξαρτήματα για την αγορά γενικά και είσαστε και τεχνικές υπηρεσίες. Η εταιρεία σας έχει λοιπόν πολλά τμήματα. Είναι σωστό αυτό εξαρτήματα ε, και τεχνικές υπηρεσίες ε, και εξαρτήματα για τους κατασκευαστές. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ε, το λέμε Original Equipment Business ή After Market Business. Ακριβώς όπως τα είπατε είναι αυτό που περιλαμβάνει το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο. Οι τεχνικές σας υπηρεσίες και αυτοί που κατασκευάζουν τα πρωτότυπα εξαρτήματα για τους κατασκευαστές έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ε, συμβουλές να δώσουν όταν, αυτό που, όταν κατασκευάζεται εξαρτήματα για τη Volkswagen παραδείγματος χάρη. Νομικές συμβουλές, τεχνικές συμβουλές Also bei den Τεχνικές υπηρεσίες λειτουργούν ω εξή. Όταν θέλουμε να παραδώσουμε ένα σύστημα, ένα σύστημα ψεκασμού για παράδειγμα, τότε αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Χρειάζεται λοιπόν ε, να καθοδηγήσουμε, να καταρτήσουμε τον πελάτη πάνω σε αυτό, να, το, να τον ενημερώσουμε. Ε, να, γιατί Κάθε κινητήρας είναι διαφορετικός. Αυτό το σύστημα έγχυσης πρέπει να προσαρμοστεί στον συγκεκριμένο κινητήρα και επίσης να λειτουργήσει σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Χρειάζεται λοιπόν ε, αυτή η τεχνική υπηρεσία, έτσι όπως τη λέμε, η οποία επικοινωνεί με τον πελάτη και τον συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ε, διαδικασίας. Ε, Τώρα, νομικά δεν ξέρω ακριβώ πώ έχουν τα πράγματα. Τεχνικά ε, μπορώ να σα απαντήσω και ναι, αυτή είναι η αρχή λειτουργία. Ναι. Ε, ε, εργάζομαι για ένα νέο τύπο νομοθεσία. για να δούμε την σχέση ανάμεσα στους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού και τις τεχνικές υπηρεσίες. Η Volkswagen χρησιμοποιεί τις τεχνικές σας υπηρεσίες στην δική της δουλειά. Ή και αυτό είναι απόρριτο. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι εμπιστευτικό αλλά να διευκρινίσω αυτά που είπε ο συνάδελφο. Κατάλαβα τι εννοείται με τεχνικέ υπηρεσίε. Τεχνικέ υπηρεσίε δηλαδή οι οποίε συνεργάζονται με τον κατασκευαστή όταν αυτό προετοιμάζει τη διαδικασία έγκριση τύπου. Αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που είπε ο κύριο Κρούγκερ. Η τεχνική υπηρεσία, έτσι όπω την εννοούμε εμεί, είναι μια υπηρεσία η οποία τα, τα εξαρτήματα τα δικά μα τα φροντίζει να ταιριάζουν με τα εξαρτήματα των άλλων προμηθευτών και του κατασκευαστή. Η τεχνική τώρα υπηρεσία με την έννοια της ε, στήριξης του κατασκευαστή για την έγκριση τύπου είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε. Εμείς δεν ε, ασχολούμαστε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ε, διευκρίνηση. Καταλάβατε, ικανοποιήθηκατε από την απάντηση. Κύριε Σούλτσα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για σας να έρθετε εδώ. Θέλετε από τη μία να απαντήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείτε, αλλά από την άλλη έχετε και αυτούς τους περιορισμούς που δεν σας επιτρέπουν να το κάνετε. Είμαι και εγώ ίδιος μηχανικός και πρέπει θέλω να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις το έχω δει και εγώ ίδιος από του ε, μικρούς προμηθευτές μέχρι έναν τεράστιο κολοσσό όπως εσείς. Ο κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού ξέρει ακριβώς τι παίρνει σε κάθε στάδιο της ε, διαδικασίας και πρέπει να το κάνει αυτό γιατί θέλουν να ξέρουν τι, τι μπαίνει στα αυτοκίνητά του, στα προϊόντα τους. Εσείς σε μία σε έναν πελάτη όπως η Volkswagen. Τι ακριβώς κάνετε. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή για έναν τόσο μεγάλο πελάτη όπως η Volkswagen να μην ξέρετε 100% τι ακριβώς ε, θα μπει στο αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, με το 100% είναι κάπως προβληματικό. Ναι, επί της ουσίας έχετε δίκιο. Η κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού πρέπει να ξέρει τι ακριβώς παίρνει για να ξέρει και αν έχει νόημα να τα συναρμολογήσει, να συνδυαστούν αυτά. Ναι, ωραία. Να κρατούσε κάτι άλλο τέλο πάντων. Ε, Μα είπατε ότι στι Βρυξέλλε. Έτσι όπως διεξάγονται οι συζητήσεις, ε, είστε κι εσείς μέρος αυτών των συζητήσεων. Στο παρελθόν όμως υπήρξε ποτέ κάποια περίπτωση για την οποία θα λέγατε ότι σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών έχει υπάρξει κάποια απόφαση που να είναι τόσο φιλόδοξη έτσι ώστε στην Ευρώπη να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν, δεν μιλάω για την Αμερική εδώ, για την Ευρώπη μιλάω. Έχει υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απόφαση νομοθετική που να, ε, είναι υπερβο, να έχει υπερβολικές απαιτήσει. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία τεχνική εταιρεία και έργο μας είναι ακριβώς να αξιολογήσουμε το αν κάτι είναι, ε, μπορεί να εφαρμοστεί, αν κάτι είναι εφικτό οικονομικά είτε και τεχνικά. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι σε μία περίπτωση μας είχαν ε, μετά το Σεπτέμβριο του του 2015 είχε γίνει μια πρόταση, η πρώτη πρόταση της Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2015 για τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και οι τιμές αυτές ήταν πραγματικά φιλόδοξες, υπερβολικά φιλόδοξες. Τότε είχαμε διεξαγάγει μια τεχνική ανάλυση για το τι ακριβώς θα ε, σήμαινε ε, αυτό εάν αυτή η νομοθεσία εφαρμοζόταν από το 2017 και μετά. Τι θα έκανε στην αγορά, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Και κάναμε λοιπόν τις δικές μας εκτιμήσεις για τους για το πόσο φυκτό είναι αυτό. Κάναμε και τις δικές μας εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην πολιτική, στην αγορά, στην, ε, στον ε, ε, στόλο μιας, ενός κατασκευαστή αυτοκινήτου. Πόσους, πόσοι περιορισμοί υπάρχουν. Και μία λοιπόν από αυτές τις συνέπειες θα μπορούσε να είναι ότι στα πρώτα στάδια της ε, χρήσης του τεστ σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, δεν ξέρουμε, ε, μάλλον τα αυτοκίνητα diesel θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσουν αυτά τα τεστ. Και αυτό λοιπόν θα οδηγούσε σε οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες φυσικά συνδέονται και με άλλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν ναι, όσον αφορά αυτό ναι. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ερτούγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Μπίζενπαχ, Δόκτωρ Κρούγκερ, καταρχάς να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ που ε, ήρθατε εδώ ένας τόσο μεγάλος ε, γερμανικός ε, επιχειρηματικός κολοσσός. Τώρα, σας λέει κάτι το χέρι Αυτά τα ονόματα δεν σας λένε τίποτα. Όχι. Ναι, ωραία, να σας βοηθήσω. Αυτά, αυτά τα δύο ονόματα είναι αυτοί που υπέγραψαν αυτήν την ε, δήλωση αποποίησης ευθύνης. Σας λέει τίποτα αυτό. Ε, δεν μπορώ να στο σχολιάσω. Δεν ξέρω από πού έχετε αυτή την πληροφορία. Εγώ δεν την έχω. Ε, δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν θα το κάνω. δεν πειράζει, δεν πειράζει, λέει ο κ. Σερτούγκ. Μια άλλη ερώτηση. Στην εταιρεία σας υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι προστατεύουν όσους καταγγέλουν παρατυπίες. Τι εννοείται δηλαδή, whistleblower εννοείται δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει στην εισαγγελία ή σε κάποια εξωτερική αρχή και θα καταγγείλει κάτι, έτσι δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιος κάποια εσωτερική τέτοια υπηρεσία, είτε που προστατεύει είτε που δεν προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω μία απάντηση γιατί δεν γνωρίζω. Δείξτε κατανόηση παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Uh, δεν είμαι συνηθισμένη στο να ολοκληρώνετε τόσο γρήγορα. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, κύριους Κρούγκερ και Μπίζενμπαχ για το χρόνο που μας αφιερώνουν σήμερα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να μου δώσετε διευκρινήσεις είναι το εξής. Εδώ συζητάμε το ε, θέμα δημοσιοποίησης ε, στοιχείων εδώ και αρκετό καιρό. Μπορείτε εσείς να μου απαντήσετε ως τεχνικός ε, εμπειρογνώμονας για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όταν γίνει υποχρεωτικός ο ε, υποχρεωτική δημοσιοποίηση ε, των στοιχείων. για αυτά τις, αυτούς τους μηχανισμούς αλλίως είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, τι, τι γίνεται ακριβώς στην πράξη. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει με του... όταν συνεργάζεται με μια τόσο μεγάλη εταιρεία όπως η ε, Volkswagen, τι γίνεται στην πράξη. Ωραία, ας αρχίσουμε έτσι. Ε, κώδικας τέλο πάντων στον οποίο αναφέρεται είναι μεγάλος. Ο κώδικας μπορεί να αποτελείται από χιλιάδες, εκατομμύρια χαρακτήρες. Τώρα η λειτουργία του είναι περίπλοκη. Αν κάποιος τώρα σε αυτόν τον κώδικα, ας πούμε μια τεχνική υπηρεσία προσπαθήσει να τον αξιολογήσει, φανταστείτε είναι τεράστιο το έργο, είναι σχεδόν άλλη το αυτό. πρέπει όταν λοιπόν μιλάμε για αυτήν την στρατηγική Based Emission Strategy, Auxiliary Emission Strategy και μας ε, ζητείτε να περιγράψουμε ακριβώς πώς ε, λειτουργεί αυτό το λογισμικό, ακριβώς πώς μειώνονται οι εκπομπές, με ποιον τρόπο αυτό είναι τεράστια δουλειά και, αλλά πιστεύω πως ε, πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άλλον τρόπο περιγραφής του ε, συστήματος αυτού. Λοιπόν, να, εγώ να σας πω για το ότι θεωρώ ότι η δημοσιοποίηση και η διαφάνεια του λογισμικού διαχείρισης εκπομπών ενός οχήματος στα πλαίσια της έγκρισης τύπου είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία την οποία δεν είχαμε στην Ευρώπη ή την έχουν στι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι κάτι που θεωρούμε πως θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, στην Ευρώπη, στην διαδικασία έγκρισης. Αυτό πιστεύω πως είναι στο σωστό. Να ρωτήσω και κάτι παραπάνω. Ναι, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, με βοήθηση η απάντησή σας. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος έχει την τελική ε, ευθύνη, ποιος κάνει τον τελικό έλεγχο πριν βγει ένα αυτοκίνητο στην αγορά. Ε, συμμετέχετε ω boss στη διαδικασία ή είναι ο κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού. Αυτό ακριβώ που είπατε, ο κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού κάνει του τελικού ελέγχους πριν διατεθεί ένα όχημα στην αγορά. Και για το λογισμικό να σα πω, Εμεί δεν αναπτύσσουμε λογισμικό, δεν γράφουμε κόμματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, εγώ άκουσα τις ε, δηλώσεις ε, που είπε ο μιλητής και θέλω να ρωτήσω το εξή, Στην πλατφόρμα που περιγράψατε με το Excel μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαδικασίες που είναι on ή off όταν το χάρη είναι στην εξέδρα τη δυναμομετρική το αυτοκίνητο, δηλαδή εσείς έχετε ένα κατάλογο ε, χάρη των λειτουργιών που μπορεί να είναι on ή off όταν είναι στην εξέδρα το αυτοκίνητο, έχετε αυτόν τον κατάλογο που αφορά το software, το λογισμικό. Δεν είμαι πολύ το σίγουρος για το τι εννοείται. Μας είπατε πολλές φορές, μας αναφέρατε καταλόγους, λίστες. Τι εννοείται δηλαδή, checklist, έναν κατάλογο με πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα φύλλο Excel και εγώ ε, θα ήθελα να αναφερθώ πριν του χάρη στο λογισμικό. Εκεί στο λογισμικό προστίθενται διάφορες διαδικασίες, ε, διάφορες φόρμουλες, διάφοροι τύποι. Εσείς εξήγησατε πάρα πολύ καλά το θέμα των τροχών, παραδείγματος χάρη και είπατε ότι όταν είναι στην εξέδρα το αυτοκίνητο δεν είναι το ίδιο όταν τρέχει στον δρόμο αλλά υποθέτω ότι κάθε κατασκευαστής σας ζητά κάποια πράγματα και να υπάρχει ένας διακόπτης on-off όταν πάει το αυτοκίνητο στη δυναμητρική εξέτα. Δηλαδή, εσείς έχετε ένα τέτοιο κατάλογο και μάλιστα μπορείτε να το δώσετε και ως απόρριτο έγγραφο στο Ε, όταν διαπιστώνονται αυτές οι παρεμβάσεις στο σύστημα εκπομπών πρέπει να, ε, να υπάρχει ενημέρωση, πρέπει να κοινοποιούνται. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβολές ε, στο σύστημα, στο λογισμικό εκπομπών που επιτρέπονται επιτρέπονται όταν ε, πρόκειται για κάποια, ε, για κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα θέματα ασφαλείας. Τώρα, το αν αυτά δημοσιεύονται, το αν, είναι, ε, αν αποτελούν εμπορικό μυστικό, αυτό εξαρτάται από το πώς ερμηνεύεται και πώς εφαρμόζεται ο κάθε κανονισμός. Αλλά υπάρχει τέτοιο κατάλογος, γιατί υπήρχαν ε, και άλλε ερωτήσει από ήταν ε, καλό να το ελέγξετε σε ιστορικό επίπεδο, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. πολύ σύντομα, παρακαλώ. Στην περίπτωση των ε, ευθυνών τι οποίε τις οποίες έχει ο κατασκευαστής, εσείς γνωρίζετε αν εσείς ε, αναλύσετε σε κάθε έναν από, το πελάτης, από τους πελάτες σας ε, τις ε, ευθύνες που υπήρχαν, αλλά και κάτι ακόμα, εσείς έχετε περιθώριο και ποιο περιθώριο έχετε να αλλάξετε την παραγγελία του πελάτη ανάλογα με τις νομικές ευθύνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπάρχει κάποια νομική βάση που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Ähm, δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση γιατί αναφέρεστε στις ε, επαγγελματικές σχέσεις ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες μας και αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, αποτελεί μέρος ε, του εμπορικού απορρίτου. Καταλάβετε με. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ε, περιστρέφονται γύρω από τεχνικά θέματα. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να αναφέρω μερικά θέματα ηθικά. Το λογισμικό σας χρησιμοποιείτε ως ε, σύστημα παραποίησης. Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν προσπαθήσατε να προειδοποιήσετε τους καταναλωτές κατά κάποιο τρόπο αν προειδοποιείτε ε, τους κατασκευαστές και θα έπρεπε και αρχές όπως η Κομισιόν να κάνουν το ίδιο πράγματα. Ξέρω ότι κερδίζετε πάρα πολλά χρήματα, αλλά αναδρομικά πόσο δαπανηρό ήταν αυτό για σας τόσο σε χρήμα όσο και σε φήμη αυτό το σκάνδαλο. ich glaube nicht, dass es dann... Δεν Νομίζω πω ισχύει κατά σας είπα, πως και από την πλευρά της βιομηχανία και από την πλευρά του νομοθέτη ήταν σαφές και γνωστό από την αρχή ότι υπήρχαν διαφορέ ανάμεσα στα αποτελέσματα των τεστ ε, σε εργαστηριακέ συνθήκε και στις ε, πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Οι, προδιαγραφ... οι τεχνικές προδιαγραφές, ε, σας είπα, σε γενικές γραμμές όσο που το πλήστο πληρούνται έτσι ώστε η επόμενη γενιά δίζελ να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα όρια εκπομπών. Ε, υπήρξε λοιπόν αυτή η προσμονή για βελτίωση της τεχνολογίας τώρα. Σίγουρα υπάρχουν οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, πρέπει να, τηρεί, να, είναι καθόλου νόμιμες. Αυτό ισχύει και για εμάς φυσικά. Τώρα, εάν διαπιστωθεί ότι έγιναν ενέργειες που δεν ακολουθούσαν την νόμιμη οδό, αυτό είναι κάτι που πλήττει όλο τον κλάδο, όχι μόνο εμάς συγκεκριμένα. Διότι δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος από μας. Η δική μας επιχείρηση, όπως ε, σας είπα, ενδιαφέρεται να ε, διαλευκανθεί όλη η υπόθεση και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Αλλά μόνο όταν έχουμε το αποτέλεσμα στα χέρια μας ε, θα μπορώ να σας πω περισσότερα. Το αποτέλεσμα των ερευνών. Um, um, Ευχαριστώ. Ίσως μια τελική ερώτηση διότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά αυτοκίνητα είναι στο δρόμο και ξέρουμε ότι με ανάκληση και με επαναρρύθμιση του λογισμικού ήδη τα αυτοκίνητα αυτά θα έχουν λιγότερες εκπομπές. Ίσως λοιπόν η πραγματική ερώτηση είναι οι κατασκευαστές πρωτοτύπου εξοπλισμού μπορούν να κάνουν αυτή τη νέα ρύθμιση ε, για να μειώσουν ε, τις ε, εκπομπές και να επηρεάσουν το σύστημα παραποίησης. Μπορεί οι κατασκευαστές να κάνουν αυτή την αλλαγή ή είναι η δική σας σύμπραξη απαραίτητη. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού. Αυτός έχει και την ευθύνη. Ε, αυτός πρέπει να ε, το κάνει. Τώρα όμως όποια αλλαγή τροποποίηση γίνει στον ε, μηχανισμό ελέγχου κινητήρα αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με εμάς φυσικά γιατί εμείς έχουμε κατασκευάσει ένα κομμάτι αυτού του κινητήρα μετά από 22 λεπτά σβήνουν ορισμένα συστήματα. Αν θέλετε νέα ρύθμιση, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια ή όχι. Wenn man mal zum Beispiel an so Ωραία, α δούμε έναν χρόνο διακόπτη για παράδειγμα. Τότε ο κατασκευαστή του πρωτότυπου εξοπλισμού πρέπει να ε, διαπιστώσει αν αυτή η λειτουργία γίνεται να ε, αλλάξει. Αν μπορεί ο χρονοδιακόπτη να ε, τροποποιηθεί. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Αυτό είναι ένα μηχανισμός προστασίας. Τώρα, Μόνο λοιπόν ο κατασκευαστής του πρωτότυπου εξοπλισμού μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές. Εμείς δεν μπορούμε σαν ε, boss να ε, κάνουμε κάτι τέτοιο, να παρέμβουμε σε αυτό. Και μία παρατήρηση από μένα. Σε, στις ε, χώρες της Ευρώπης υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις προϋποθέσεις και την νομοθεσία για την αλλαγή των, του λογισμικού, αλλαγή του λογισμικού κινητήρα μέχρι ένα σημείο αυτές οι τροποποιήσεις είναι αποδεκτές όπως σας είπα και πολλές φορές γίνονται δεκτές από τις ε, αρχές ελέγχου ως ε, απόλυτα φυσιολογικό. Μια ερώτηση ε, σχετικά με την παρακολούθηση της αγοράς για οποιαδήποτε προϊόν η αρχή παρακολούθησης της αγοράς πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντα. Ε, νομίζω ότι τα αυτοκίνητα πρόκειται περισσότερο για λογισμικό παρά για μηχανική. Πώς οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν ότι γνωρίζουν επακριβώς τι κάνει το λογισμικό σας και αν δεν χρησιμοποιείτε για να παρακάμψει τον νόμο. Οι λογικές συνέπειες θα είναι και οι ερωτήσεις είναι όταν οι αρχές έγκρισης τύπου οχήματος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πηγή ε, του λογισμικού. Έτσι δεν είναι. Ο συνάδελφος απάντησε για το τελευταίο σας ερώτημα τώρα, για την πρώτη ερώτηση. Ε, αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσετε στους αρμόδιους, αυτούς που είναι αρμόδιοι για την έγκριση. Εμείς πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαδικασία έγκρισης αφορά α, τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ε, περισσότερο. Είναι κάτι ανάμεσα σε αυτούς και στις αρχές έγκρισης. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Yes, I, do Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα συζητούμε τώρα μια νέα ε, νομοθεσία για την έγκριση τύπου ε, και θα θέλαμε να έχουμε τις απόψεις σας, τις απόψεις κάποιου που ασχολείται με το λογισμικό. Είσαστε από, ε, τα σημαντικότερα μέρη της διαδικασίας κατασκευής αυτοκινήτων. Μήπως πρέπει να, να αλλάξουμε το σύστημα έγκρισης τύπου, τη διαδικασία ως προς το θέμα αυτό. Τι πιστεύετε. Ναι, αλλά όπως είπα και πριν, έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή με την ε, τροποποίηση, την ε, επικαιροποίηση της, της οδηγίας τον Ιούλιο, όπου το η βασική στρατηγική εκπομπών, το Basic Emission Strategy, έχει οριστεί. Έχει οριστεί επίσης και μία ε, βοηθητική στρατηγική για τις εκπομπές, Auxiliary Emission Strategy. Αυτό ε, φυσικά χρειάζεται και ε, προϋποθέτει μάλλον να η έγκριση τύπου να, να γίνεται με διαφάνεια. Αναμένεται ακόμα η απόφαση του ε, Κοινοβουλίου, δεν ξέρω εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά νομίζω πως σε γενικές γραμμές πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, μέχρι τώρα. Να πω κι εγώ κάτι, να προσθέσω κι εγώ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Ε, ε, αλλά όσον αφορά το λογισμικό, είμαστε έμεσα εμπλεκομένοι, δεν μας αφορά άμεσα. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει κάποια σύγχυση εδώ, γιατί πάρα πολλοί πρέπει να φύγουν για την Ολομέλεια. Ε, χαίρομαι που έχω λίγη, λίγο χρόνο για να επανέλθω στο θέμα των τεχνικών υπηρεσιών. Στον ιστότοπο λέει ότι η Bosch ε, παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την έγκριση τύπου. Το κάνετε αυτό στην εταιρεία σας και είπατε ότι η Volkswagen δεν χρησιμοποιεί τις τεχνικές σας υπηρεσίες, αλλά αλλά η ερώτησή μου είναι, εσείς μέσα, μέσα στην Bosch, στην εταιρεία σας, χρησιμοποιείτε την γνώση που έχετε από τις τεχνικές υπηρεσίες για να βοηθήσετε τα άτομα που εργάζονται με πρωτότυπα εξαρτήματα μέρη της Volkswagen υπάρχει κάποια ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις ε, τεχνικές υπηρεσίες και ξέρουν τι απαιτείται από την νομοθεσία και αυτούς που κατασκευάζουν εξαρτήματα για τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού. Also, ich will nochmal die äh, Έχουμε συζητήσει τη διαφορά που υπάρχει. Από τη μία λοιπόν υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες όπως σας είπα οι οποίες συνεργάζονται με τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού για τη διαδικασία έγκρισης. Αυτή, ε, αυτή η διαδικασία εποπτεύεται και από τεχνικούς, ε, τεχνικές ενώσεις ε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία. Οι τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ε, αναφέρθηκαν από εμά, από τον κύριο Κρούγκερ, έχουν να κάνουν με την δημιουργία, με το σχεδιασμό ενός προϊόντος, με την ε, παράδοση ενός προϊόντος το οποίο πρέπει να ε, ταιριάζει με τις συγκεκριμένους κινητήρες. Νομίζω, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Ίσως, αλλά νομίζω καλό είναι να τα διαχωρίσουμε στο μέλλον. Μια πιο γενική ερώτηση τώρα. Θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο στην ομοθεσία για την έγκριση τύπου να έχουμε ένα σύστημα για τους καταγγέλλοντες, για τους whistleblowers. Αν κάποιος δηλαδή γνωρίζει κάτι και μιλώ γενικά, θα μπορούσε να δίνει πληροφορίες στις αρχές σχετικά. Νομίζετε ότι θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο ως μια εταιρεία που προμηθεύει τους κατασκευαστές πρώτα του εξοπλισμού με εξαρτήματα. Äh, Δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Ε, ε, τουλάχιστον εμείς Θεωρούμε πως σε ό,τι αφορά τις, ε, τα όρια εκπομπών, την έγκριση τύπου, τις ε, προϋποθέσεις για τα επιμέρους εξαρτήματα υπάρχουν συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένα όρια αναφέρεται ρητά από την νομοθεσία. Τώρα εμείς θεωρούμε πως τα νέα στοιχεία για την έγκριση τύπου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δηλαδή τα τεστ στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη για παράδειγμα, ζητείται μια τέτοια εναρμόνιση της νομοθεσίας για ε, το θέμα αυτό, για τις εκπομπές. Ε, υπάρχει επιθυμία να ε, διαμορφωθεί κοινή νομοθεσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη παγκόσμια. Τώρα, ε, η βιομηχανία και οι προμηθευτές συγκεκριμένα ε, ιδανικό θα ήταν ε, κατά αυτούς, κατά εμάς δηλαδή, να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές παγκοσμίω. Ε, να υπάρχουν δηλαδή, ή να υπάρχει διανομοθεσία να υπάρχει το ίδιο πλαίσιο για αυτό. Βέβαια, πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στην νομοθεσία ανά τον κόσμο και σε αυτό προσπαθούμε να προσαρμοστούμε εξάλλου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνουμε την ακρόασή μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του κύριου Κρυγκίρ και Μπίσενπαχ. Σημειώσατε ότι υπάρχει κάποια σύγχυση και απογοήτευση για το ότι δεν μπορείτε να μα απαντήσετε σε όλα. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που έχουν παραμείνει. Θα υπάρξουν και κάποιες γραπτές ερωτήσεις, όπως συμφωνήσαμε και από την κυρία Κάντεμπαχ. Αν έχετε ερώτηση, στείλτε τη γραπτός. Και δεύτερον, αν είναι δυνατόν και έχετε κάποια ένδειξη για το πότε θα ολοκληρωθεί η εσωτερική σας έρευνα και ιδίω τα σημεία που μπορούν να δημοσιευτούν, θα ενδιαφερόμασταν πάρα πολύ να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε εδώ στο Στρασβούργο, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω δύο ανακοινώσεις. Ε, καταρχήν ε, η απόφαση της συνάντησης των συντονιστών της 1 Σεπτεμβρίου είναι στο φακελό σας και αν δεν έχετε αντίρρηση θα υιοθετηθεί. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 26 Σεπτεμβρίου είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα συναντήσουμε τις Αμερικανικές Αρχές, την EPA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή ψηφοφορία και καλή επιστροφή.